The Good afternoon, colleagues. Um, welcome to the... Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην απογευματινή συνεδρίαση. Τα χθεσινά πρακτικά είναι διαθέσιμα και αν δεν υπάρχουν σχόλια... Συγγνώμη, παρακαλώ, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να